Good morning, Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου. Ελπίζω να μην διαμαρτυρηθεί κάποιος με αυτά τα οποία έχουμε στη μερίσια διάταξη αυτονόητα. Δεν έχω άλλες ανακοινώσεις να κάνω. Μπορούμε να περάσουμε απευθείας στο κύριο θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης. Η απαλλαγή για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για το 2016 και με ευρωπαϊκό τρόπο θα έλεγα. Έχουμε τρεις σχολιαστές, τον κύριο Ρούσο από το ελεγκτικό συνεδρίο, ο οποίος πρώτος θα πάρει το λόγο. Ε, μετά έχουμε την Αντιπρόεδρο Μογκερίνη. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να συντονιστείτε με τις δικές μας ε, επιθυμίες ε, και χρονοδιαγράμματα. Και έχουμε και τον εισηγητή, ο οποίος είναι Ιταλός. Τώρα δεν είναι μόνο Ιταλός ο εισηγητής, αλλά και η κυρία Μογκερίνη και ο κύριος Ρούσο και μετά μπορούμε να περάσουμε σε σχόλια και ερωτήσεις. Έχουμε 90 λεπτά. Στην ουσία μπορούμε να παίξουμε ένα αγώνα ποδοσφαίρου. Ξέρω ότι πολλές φορές όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου θέλουν να βάλουν γκολ, οπότε θα πρέπει να φροντίζετε το χρόνο που θα ομιλείτε. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας τον λόγο στον κύριο Ρούσο, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Rapporteur, members of the Committee on Budgetary Control, Είμαι εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να παρουσιάσω την αξιολόγηση για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Είναι θετική η αξιολόγηση και τα διοικητικά θέματα και οι πληρωμές δεν επηρεάζονται από προβλήματα πρακτικά. Η αξιολόγηση έγινε μέσα από 100 περιπτώσεις τις οποίες εξετάσαμε. Βρήκαμε 5 από αυτές να έχουν κάποια λάθη, ιδιαίτερα στις προμήθειες. Αντίστοιχα με αυτά τα οποία είχαμε διαπιστώσει και τον προηγούμενο χρόνο, το 2015. Οι διαδικασίες προμηθειών δεν είναι οι κατάλληλες μερικές φορές, Υπάρχουν ελλείψεις τεκμηρίων σχετικά με κάποια βήματα της διαδικασίας και ε, δεν υπήρξε σε ορισμένες περιπτώσεις σεβασμός των προθεσμιών. Αξιολογήσαμε περαιτέρω ότι σε σχέση με τις συστάσεις τις οποίες είχαμε κάνει το 2013 για τη διαχείριση των οικογενειακών ε, επιδομάτων ε, να είναι σωστοί και να είναι επιμέρους η εφαρμογή των συστάσεων σε σχέση με τις διαδικασίες προμηθειών. Και αυτό το ε, ανέφερα ε, ίσχυε και το 2015 ισχύει και φέτος. Φέτος εννοώ για το 2016. Όπως ε, υπόθηκε και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής, το ελεγκτικό συνεδρίο εξέτασε και την εφαρμογή του στόχου της μείωσης του προσωπικού κατά 5% όπως είχε αποφασιστεί από τις αρχές επί του προϋπολογισμού του 13. Οι αξιολογήσεις μας περιλαμβάνονται στην, πρόσφατα, ε, στην πρόσφατη έκθεση την οποία, η οποία κυκλοφόρησε. Υπάρχει συμβατότητα με τους στόχους. Βέβαια η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, ξεκίνησε τη διαδικασία μείωσης του προσωπικού της ένα χρόνο αργότερα, οπότε η τελική αξιολόγηση θα γίνει στο τέλος του 2016. Παράλληλα, δημοσιεύσαμε και την τομεακή μας έκθεση υπαριθμών 7 το 15 για την χρήση των κτηρίων της υπηρεσίας αυτής στον κόσμο. Γενικά τα κτίρια καλύπτουν τις ανάγκες των αντιπροσωπιών, αλλά μερικές φορές δεν διασφαλίζουν το καλύτερο λόγο, την καλύτερη σχέση ανάμεσα στο κόστος και στα όφελος ε, μέσω της χρήσης τους. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας, κυρία Αντιπρόεδρε και κύριε Πρόεδρε, για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μογκερίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, διότι... Εσύ δεν μπόρεσα να παραστώ στη συνεδρίαση που είχαμε προβλέψει να έχουμε στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Ήμουν και εγώ θύμα τη γρήπη τέτοια εποχή. Χαίρομαι που σήμερα έχουμε το περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό που για μένα είναι σημαντικότατο βήμα όσον αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής ε, δράσης. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας εσάς κύριε Πρόεδρε, τον εισηγητή, προφανώς το έργο που επετελέστη αυτές τις εβδομάδες και μήνες ήταν σημαντικό, ευχαριστώ. Θέλω να συζητήσουμε μαζί πώς η υπηρεσία μας μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη. Είναι η τέταρτη φορά που μιλώ σε εσά σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτά τα τρία χρόνια είδαμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να εξελίσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει συνεχώς να προσαρμόζουμε τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίου εργαζόμαστε, ούτως ώστε να προσαρμοζόμαστε ε, σε αυτό τον εντυπωσιακό ρυθμό. Υπάρχει νέα ζήτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται να είναι ισχυρός ε, φορέας στο προσκήνιο το Διεθνέ της Πολιτική. Είμαστε όλο και πιο απαραίτητοι εταίροι στα σημαντικά ζητήματα της εποχής μας και αντιμετωπίζοντα προβλήματα αυξανόμενα στο περιβάλλον καθημερινά βλέπω στη δουλειά μου ότι υπάρχει μεγαλύτερη επίγνωση όσον αφορά την ανάγκη για ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση στον κόσμο, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε όλο τον κόσμο, σε πολλά μέτωπα. Αυτό αληθεύει ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στα κράτη-μέλη. Σκεφτείτε το θέμα της μετανάστευσης. Πριν από τρία χρόνια η μετανάστευση δεν ήταν ακόμα τμήμα του έργου του εξωτερικού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, δεν είναι και στο έργο τη υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και τώρα η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική βασίζεται πολύ στην δουλειά που κάνουμε, στη συνεργασία με του εταίρου μα στον κόσμο, με την υπατερμοστία για τους πρόσφυγε του ΟΗΕ, με τον ΟΗΕ και στο, με το, το έργο των κρατών μελών κατά πολύ εξαρτάται από την κοινή μα εξωτερική δράση για τα σύμφωνα μεταναστεύσεως, τα καταπαστεύματά μας, για τις, στις αποστολές ε, στρατιωτικού τομέα, ιδιωτικού τομέα συνεργασία από την Αφρικανική Ένωση και με τον ΟΗΕ και μέσω των συμφωνιών που έχουμε με μας στον κόσμο από το Πακιστάν μέχρι άλλες χώρες της Ασίας, για να μην αναφέρω την Αφρική. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα το πώς οι προσδοκίες και το πεδίο δράσης μας έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια. Επίσης υπάρχει μεγαλύτερη επίγνωση του ρόλου μας εκτός Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Έχουμε γίνει σημείο αναφορά όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην περιοχή μα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο από την Νότια Αμερική μέχρι την Άπο Ανατολή, από την Αφρική μέχρι την Αρκτική. Εάν δείτε μία από τι που έχουμε ω Ένωση και σαν Κοινοβούλιο, όπω γνωρίζω, δηλαδή την ενίσχυση και την επιβίωση καμιά φορά των, του πολυμερού συστήματο που έχει ενταχθεί στο σύστημα του ΙΕ, Παίρνετε την οικογένεια του ΟΗΕ και βλέπετε ότι προσβλέπει σε εμά ο ΟΗΕ για υποστήριξη ε, για θέματα όπω είναι η αλλαγή του κλίματο, όπω είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ειρηνευτικέ ε, αποστολέ. Κύριε, όπω ξέρετε, ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Κουτιέρε, έχει πολύ ε, φιλόδοξα σχέδια τη μεταρρύθμιση του οργανισμού και βασίζεται σε εμά για να το πραγματοποιήσει αυτό και να τον υποστηρίξουμε σε διάφορου τομεί. Και για να συνεχίσουμε με κανένα δύο παραδείγματα, θα γνωρίζετε πώ είμαστε στο κέντρο των προσπάθειών για τη διατήρηση συμφωνία με το Ιράν, πόσο σημαντική έχουμε γίνει όσον αφορά τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη. Συνεργαζόμαστε με του εταίρου μα στο Κουαρτέτο και με την Αραβική ε, τον Αραβικό Σύνδεσμο και είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Νετανιάχου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό. Ή σκεφτείτε τη δουλειά που κάνουμε στα πλαίσια διαδικασία των Βρυξελών για τη Συρία και για του Σύρου και εντό τη χώρα και εκτό τη χώρα και τις προσπάθειες που καταβάλουμε στο Ιράκ, όπου ήδη έχουμε κάνει μια αποστολή πολιτική για να υποστηρίξουμε διάφορες μεταρρυθμίσεις στη χώρα σε κρίσιμη εποχή και εκεί θα συμπροεδρεύουμε τις διασκέψει των οικοδομήσεων σε μερικές εβδομάδες στο Κουβέιτ. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει που ανέφερα, σαν παραδείγματα, είναι παραδείγματα που θα μπορούσα να συνεχίσω να πάμε από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τη Χιλή, Καναδά, η Ιαπωνία. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει ο ρόλο μα είναι μοναδικό όσον αφορά την ε, ισχύ που προωθούμε, δημιουργούμε κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ των ε, τέρων μα όσον αφορά τι ανθρωπιστικέ προσπάθειε, τι καλέ σχέσει με του πιο σημαντικού φορεί και προφανώ όλα αυτά εδράζονται επί των κοινών ευρωπαϊκών μα αξιών. Θα ήθελα να πω το προφανέ ότι όλο και περισσότερο είμαστε ένα σημείο αναφορά και στη δική μα Ήπειρο με εκείνου εταίρου οι οποίοι δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι Ευρωπαίοι. Καταρχάς και πρωτίστως είμαστε σημείο αναφοράς για τους ανατολικούς μας εταίρους. Αυτό είναι το μήνυμα που όλο και περισσότερο ακούω από αυτούς, από όλους αυτούς και θέλουν περισσότερες επαφές μαζί μας, να έχουμε περισσότερο εμπόριο, να συνεργάζονται περισσότερο και να επεξεργάζονται διάφορες πτυχές της συνεργασίας μας. Προφανώς είμαστε και σημείο αναφοράς και όλο και πιο σημαντικό σημείο αναφοράς για τα Βαλκάνια διότι κάθε ένας από τους έξι εταίρους μας προσπαθεί να αλλάξει την κοινωνία του, να τη μεταμορφώσει και ακολουθούν ένα μονοπάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές φορές είπα ότι φέτος, ιδιαίτερα αυτό το εξάμεινο της Βουλγαρικής Προεδρίας, μπορεί αυτό να είναι σημείο κομβικό τους ώστε να ανοίξει το μονοπάτι του προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει μονόδρομο αυτή η πορεία και αυτό είναι προ όφελο και συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλού λόγου, όπω είναι οι οικονομικοί λόγοι και οι λόγοι ασφαλεία. και όταν έρθουμε στο θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τι βλέπω. Βλέπω ότι τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου γνωρίζουν πολύ καλά τα περιθώρια που υπάρχουν, τους χώρους που ανοίγουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε αυτή να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα περιθώρια, να τα διαρευνήσει όσον αφορά την εξωτερική δράση. Μου λέτε πάρα πολύ συχνά ότι υπάρχουν νέες ευκαιρίες που μπορούμε να κονταλευτούμε, νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ότι υπάρχουν κενά όπου εκεί θα μπορούσαμε να εισχωρήσουμε σαν δύναμη ε, ειρήνη συνεργασίας και ανθρώπινης ανάπτυξη και δεν αποτελεί σύμπτωση ότι όλοι οι δείκτες του Ευρωβαρομέτρου δείχνουν ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής σε συντριπτικό ποσοστό υποστηρίζουν περισσότερη ε, πολιτική κοινή εξωτερικής πολιτικής μάλλον και ασφαλείας την Ευρώπη, γιατί έτσι η Ευρώπη θα πετύχει πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Υπάρχει ζήτηση λοιπόν για αυξανόμενο και επεκτηνόμενο πεδίο δράση ε, σε αυτό το τομέα. Εγώ συμμερίζομαι πλήρω αυτή τη φιλοδοξία, διότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η ανθρώπινη εξέλιξη στην Ευρώπη για του πολίτε μα εξαρτάται από την κατάσταση που είναι έξω τα σύνορά μα και αυτό το είδαμε ε, σαφέστατα πρόσφατα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια όσον αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, όσον αφορά του πρόσφυγε ε, ή τι μεταστατικέ ροέ. Βλέπουμε τι διασυνέσει που υπάρχουν μεταξύ εξωτερικού χώρου και εσωτερικού χώρου τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και εδώ έρχομαι ακριβώ το βασικό σημείο τη ημερήσια διάταξη όντες ευρωβουλευτές ίσως θα ενδιαφερόσαστε όχι μόνο για τα λογιστικά θέματα, αλλά και ενδιαφέρεστε για το πολιτικό περιβάλλον που υφίσταται και αφορά τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης. Για να παίξουμε πλήρως τον ρόλο μας, θα πρέπει τα του οίκου μας να είναι τακτοποιημένα και δημοσιονομικά και συμμερίζομαι απόλυτα αυτά που συζητούσαμε πέρσι. Δηλαδή, για να ανταποκριθούμε στι αυξανόμενε προσδοκίε, χρειαζόμαστε επαρκή μέσα. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Αυτό δεν είναι το θέμα τη σημερινή συζητήσεω, βέβαια, αλλά παρακαλώ αυτό να το έχουμε υπόψη τώρα που ξεκινάμε τι συνομιλίε για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο αυξανόμενε προσδοκίε, αυξανόμενε προκλήσει, μείωση των ε, οικονομικών πόρων, θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητε και να μοιάζουν προτεραιότητε δικέ μα αυτέ των πολιτών. Ταυτόχρονα υπέχουμε καθήκον και είναι και συμφέρον μα πιστεύω να είμαστε πλήρω αξιόπιστοι, ελεγχόμενοι, διαφανεί στην καθημερινή μα δουλειά. Θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και πάντα να τηρούμε τα ύψιστα πρότυπα, διότι στη, στον τομέα τη εξωτερική ε, δράσεω η αξιοπιστία και κάποια δημοσιονομικά θέματα και ο έλεγχος και η διαφάνεια, όλα αυτά τα ζητήματα είναι η μόνη ε, δυνατή βάση για να μπορούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας. Διότι από αυτού απαιτούμε έλεγχο, διαφάνεια, λογοδοσία, διαφάνεια και αξιόπιστη δημοσιονομική συμπεριφορά. Άρα είναι ένα κομμάτι της πολιτικής. Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι της διαχείρισης. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στους ε, εταίρους μας ε, στο εξωτερικό και για τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για μένα είναι υψής της σημασίας εμείς να είμαστε 100% όπως σας είπα ελεγχόμενοι, διαφανείς, αξιόπιστοι. Λοιπόν, πολύτιμη αυτή η ευκαιρία να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι απλώς μια εξέταση της καταστάσεως, διότι δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα όπως ακούσατε που πρέπει να εξετάσουμε και οι υπηρεσίες έστειλαν απαντήσεις στις αρχικές ερωτήσεις που ετέθησαν και προφανώς είναι μαζί μου μέλη τη υπηρεσίας για να απαντήσουν σε ερωτήσεις περισσότερο τεχνικής φύσης που ίσως εγώ να μην γνωρίζω επαρκώς τις τεχνικές λεπτομέρειες για να απαντήσω, αλλά ήρθαν εδώ για να μπορέσουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που ίσως υπάρξουν. Αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι μία, δεν είναι εξετάσει αν θέλετε, δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, να ακούσουμε απόψεις, συστάσεις για το πώς η υπηρεσία μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη, πώς να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας καλύτερα και πώς μπορούμε να χειριστούμε την υπηρεσία με αποτελεσματικότερο τρόπο. Νομίζω και βλέπω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά. Όλοι θέλουμε η υπηρεσία εξωτερική δράση να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα μέσω ορθή δημοσιονομική διαχείριση και αυτό είναι ο κοινό στόχο. Όπω και σε προηγούμενα χρόνια, θεωρώ ότι αυτό είναι μια ευκαιρία για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε, να μάθουμε από την εμπειρία και να ακούσουμε τι απόψει σα επίση και να βελτιώσουμε την κατάσταση γνωρίζοντας ότι κάποια πράγματα ίσως να χρειάζονται χρόνο Ξέρετε ότι για να αλλάξει η πορεία ενός σκάφους καμιά φορά χρειάζεται χρόνος ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους, του πλοίου, αλλά είναι σημαντικό ε, να ακολουθήσουμε τη σωστή πορεία και να αρχίσουμε να βλέπουμε τις κινήσεις που κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό μετρά για μένα να ελέγξουμε και να ξαναελέγξουμε εδώ και να δούμε ότι οι αλλαγές που χρειαζόταν έχουν ξεκινήσει ήδη, έχουν δρομολογηθεί και ότι είναι σωστή η πορεία που ακολουθούμε. Η κατεύθυνση έχει κάποιου τομεί, και ανέφερα ένα-δύο, Πρέπει να επιταχύνουμε μάλιστα τι εργασίε και εκεί θα ζητήσω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να με βοηθήσει το Κοινοβούλιο στο συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, να επιταχυνθεί η εργασία μα και να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε σύντομα. Ένα παράδειγμα το οποίο βελτιώσαμε από πέρσι, από την περσινή συνομιλία μα. Και Ιδιαίτερα χάρηκα γι' αυτό και είμαι περήφανη γι' αυτό. Ο Ευρωπαίος διαμεσονοβητής σωστά είχε θέσει ένα θέμα που αφορούσε την αμοιβή των εκπαιδευμένων μας. Συνεργάζομαι μαζί μας, τους βλέπω, είμαστε σταθερά, είναι νέοι Ευρωπαίοι που ε, συμβάλλουν στην καθημερινή μας εργασία, είναι αφοσιωμένοι στην εργασία τους, δίνουν ενέργεια, έχουν δεξιότητα, δείχνουν πάθος που είναι αξιοσημείωτο και το να σπληρώνουμε αυτό ήταν ένα δικαίωμα, σωστό μάλλον πράγμα που έπρεπε να κάνουμε. Και τώρα τους προσφέρουμε και ε, υποτροφία και χαίρομαι που διαμεσομαλιδητής ε, θεωρεί ότι έχουν, έχουμε συμμορφωθεί με τις συστάσεις του. Αυτό έδειξε κάτι που μπορούσε να αλλάξει αμέσως και έγινε και είναι κάτι θετικό. Ε, και εάν άλλα θέματα είναι εύκολα να αλλάξουν, τίποτα δεν είναι εύκολα, δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, πάντα εγώ και η υπηρεσία μου θα δείτε ότι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τις δέουσες αλλαγές. Και γρήγορα και με αποφασιστικότητα. Και να δρομολογήσουμε σωστά τα δέοντα θέματα και να κινηθούμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το θέμα της υποτροφίας για τους μαθητευόμενους, πόσο κρίσιμη είναι η στήριξη των δημοσιονομικών αρχών, πώς μπορεί να βελτιώσει τις εργασίες μας και το περιβάλλον εργασίας εντός της υπηρεσίας μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Ανέφερα το περιβάλλον εργασίας για μένα, είναι κρισίμο σημασία κυρίως σε αυτή την υπηρεσία, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, εάν δεν έχει κάποιο κίνητρο, αν δεν είναι αποφασισμένος, αν δεν έχει πάθος αυτό που κάνει και αν δεν εργάζεται σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι θετικό, είναι δυσκολότατο να, να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, κυρίως ε, να έχεις κίνητρο να τα αντιμετωπίσεις, χρειάζεσαι χρόνο, να αντιμετωπίσεις περιορισμούς. Ε, λοιπόν, κατά την άποψή μου, λοιπόν, τα κίνητρα και καλό εργασιακό περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρούσο του Ελεκτικού Συνεδρίου, όχι μόνο για την παρουσία του και για τα λόγια του, αλλά και για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση για το 2016 επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό των ε, λαθών είναι κάτω από 2%, πολύ κοντά στο 0 δηλαδή, και το σύστημά μας, το σύστημα διαχείρισής μας έχει ε, επιστοποιηθεί από την Γενική Διεύθυνση του Προϋπολογισμού. Η έκθεση βέβαια αναφέρει κάποιες ανησυχίες, για παράδειγμα για διαγωνισμούς χαμηλού και μεσαίου χρηματικού επίπεδου. Ε, το, είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα για μας, στη, για τις αντιπροσωπίες μας σε τρίτες χώρες. Μην ξεχνάτε ότι ε, Πολύ συχνά οι αντιπροσωπείες μας δεν λειτουργούν σε χώρες και σε αγορές που χαρακτηρίζονται από ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για αυτές. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να τηρήσουμε τις υψηλές προδιαγραφές στους, ε, στις προκήρυξεις διαγωνισμών. Δεν λέω ότι είναι αδύνατο, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο εκτός Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης κάποιες ε, χώρες είναι πολύ ιδιαίτερες και κάποιες αγορές είναι πολύ ιδιαίτερες. Γι' αυτό το λόγο εξακολουθούμε να βελτιώνουμε την εκπαίδευση, τι ε, τις κατευθύνες γραμμές και τις διαδικασίες μας όπου είναι δυνατό. Καταλαβαίνουμε ποια είναι η πρόκληση και πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Το δίκτυό μας 140 αντιπροσωπιών είναι μοναδικό στον κόσμο είναι απαραίτητο για την εξωτερική μας πολιτική, αλλά είναι απαραίτητο όλο και περισσότερο και σε άλλες ε, σε πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να το αναπτύξουμε. Εσείς και οι συνάδελφοί σας ε, επισκέπτεστε τρίτες ε, χώρες στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, βλέπετε την κατάσταση και συχνά ε, βασίζεστε στις αντιπροσωπίες μας προκειμένου να σας συνδράμουν ε, σε συναντήσεις που έχετε. Η διατήρηση και ανάπτυξη αυτού του δικτύου έχει δημοσιονομικές συνέπειες, όπως σε όλες τις διπλωματίες στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή 820 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προπολογισμό μας σχετικά μικρός σε σχέση με τη δουλειά που κάνουν οι 7.000 άτομα, τα 7.000 άτομα του προσωπικού μας. Πολύ περισσότερο που διευρυνόμαστε όλο και περισσότερο σε ό,τι αφορά ε, το πεδίο μας, οικονομική διπλωματία, ε, ε, επενδύσεις, επενδυτές, κλιματική αλλαγή, τρομοκρατία, πολιτιστική διπλωματία. Κάθε μέρα έχουμε καινούριους κλάδους, καινούριους τομείς που ε, προστίθενται στις ε, εργασίες μας, στο πεδίο μας. Σας δώσω δύο παραδείγματα από την καθημερινή μου δουλειά. Χτες συναντήθηκα με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO και συζητούσαμε πώς επιτόπου μπορούμε, στο πεδίο δηλαδή, μπορούμε να στηρίξουμε το έργο της UNESCO για την ε, διάσωση ε, πολιτιστικής κληρονομιάς, την αντιμετώπιση ε, της αρχαιοκαπηλείας κλπ. Να για παράδειγμα ένα, ένας τρόπος ε, που διαβρύνουμε τη δράση μας. Τις προάλλες συνάντησα επίσης τους εκτελεστικούς διευθυντές των πιο σημαντικών εταιριών ε, διαστήματος διαστημικής τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ζητήσαν να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν τον προστατευτισμό που χαρακτηρίζει τον κλάδο αυτό. Με μικρά με πολύ, πολύ μικρούς προϋπολογισμούς οι αντιπροσωπείες μας κάνουν εξαιρετικό, ε, εξαιρετική δουλειά. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό και το συζητήσαμε και την περασμένη χρονιά και νομίζω ότι μπορούμε να βασίζουμε σε εσά είναι η ασφάλεια του προσωπικού μας. Αυτό το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας. Χρησιμοποίησαμε πολύ αποτελεσματικά τον προπολογισμό 2016-2017 ε, από το πακέτο ασφαλείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κοινοβούλιο που μας στήριξε με τους πρόσθετους πόρους που μας δόθηκαν. Ε, ορίσαμε, προσλάβαμε 24 πρόσθετους ε, αξιωματικούς ασφαλείας, 58 συνολικά σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή και ξεκινήσαμε και διαγωνισμό για την αγορά πρόσθετων ε, ε, τεθωρακισμένων οχημάτων. Ταυτόχρονα ε, καταρτίζουμε περισσότερο το προσωπικό μας. Ήδη ε, ε, εργάζονται σε πολύ δύσκολο περιβάλλον συχνά. Πρέπει να είμαστε παρόντες σε πολύ ευαίσθητα σημεία του πλανήτη και προφανώς αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα. Το προσωπικό μας πολύ συχνά είναι υποχρεωμένο να εργάζεται σε προβληματικό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά εργάζονται για τη δική μας ασφάλεια και ευημέρεια και θα πρέπει να φροντίζουμε και για τη δική τους ασφάλεια με επαρκείς πόρους. Όσο γινόμαστε απαραίτητος ε, εταίρους σε όλο τον κόσμο, χρειάζεται να είμαστε, όλο και περισσότερο χρειάζεται να είμαστε εκεί, να είμαστε ορατοί και να υψώνουμε τη σημαία μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά έχει ζητήσει στο παρελθόν μεγαλύτερη παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο, μεγαλύτερη ορατότητα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Προφανώς βρισκόμαστε στην εποχή της ψηφιακής διπλωματίας, οπότε όλοι μας και εγώ ίδια πρέπει να είμαστε σε επαφή με τους εταίρους, με ε, email, με whatsapp, οτιδήποτε, αλλά προφανώς η ε, προσωπική παρουσία δεν μπορεί να αποφευχθεί. Η ε, στενές επαφές ή άμεσες επαφές είναι απαραίτητες ε, για να δει κανένα και με τα μάτια του την, την πραγματική κατάσταση. Αυτό καθιστά απαραίτητο το να είμαστε εκεί. Χρειάζεται να ταξιδεύουμε πολύ συχνά, όπως οποιαδήποτε άλλη πραγματική υπηρεσία στον κόσμο, όπως και εσείς. Να εφαρμόσουμε και το έργο των άλλων ε, υπηρεσιών είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και σε αυτό το τομέα λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα ύψιστα ε, πρότυπα για την αποτελεσματικότητα διαφάνεια και να παραμείνει το κόστος στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο σε οποιαδήποτε αποστολή κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εκτελούμε αποστολές. Οι προσδοκίες όσον αφορά την εξωτερική μας πολιτική έχουν αυξηθεί. Ε, Μα ζητήθηκε από το Συμβούλιο, όπω γνωρίζετε, όμω να κάνουμε περικοπέ προσωπικού κατά 5% Ολοκληρώσαμε τέλος του περασμένου έτους, όπως είδε και το Λευκό Συνέδριο, το κάναμε αυτό. Το πετύχαμε, κάναμε τις περικοπές όσον αφορά ε, το αρχηγείο μας, αν θέλετε, περιορίζοντας τον αριθμό των ατόμων στις αντιπροσωπείες και από, θα πάει από, το, από το, την κεντρική δίκηση προς τις αποστολές θα πάνε 20 άτομα αν εγκριθεί ο προπολογισμό. Αυτό έχει εγκριθεί για το 2018 και ευχαριστώ πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την ε, ε, βοήθεια. Θα πρέπει να συνεργαζόμαστε καλύτερα και θα πρέπει να είμαστε πιο παρόντες ε, στο εξωτερικό. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε να οι ειδικοί εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Ενώσης και των προσωπικών ενταχθούν στο έργο τη υπηρεσία. Αυτό είναι κάτι που ε, σα απασχολεί όλου ιδιαίτερα, σημαντικό για εσά. Το συζητήσαμε επανειλημμένα με την επιστολή με την, με την τροποποίηση του προπολογισμού 2018 πήραμε τα αναγκαία χρήματα για την ε, ειδικό εκπρόσωπο του Αφγανιστάν να ενταχθεί στην υπηρεσία μας και βασίζομαι στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα, ώστε να πιστεί και το Συμβούλιο για την πολιτική ανάγκη για αυτή την πρωτοβουλία να συνεχιστεί. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι δύσκολο σαν εγχείρημα ε, και είμαστε μαζί στην ίδια πλευρά. Κάτι άλλο σημαντικό τομέα που επεξεργαζόμαστε είναι η ισορροπία όσον αφορά το φύλλο, γεωγραφική ε, περιοχή και ισορροπία μεταξύ εθνικών διπλωματών και μονίμων υπαλλήλων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όσο μεγαλύτερη ποικιλομορφία έχουμε στην υπηρεσία, ε, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η εξωτερική μας πολιτική, διότι έχουμε αρκετές ε, απόψεις που τις λαμβάνουμε υπόψη εξ αρχής, τις διάφορες απόψεις. Και αυτό μας βοηθά πάρα πολύ. Αυτό είναι το θετικό πρόσημο που έχουμε εμεί και δεν έχουν εθνικέ διπλωματίε. Είναι η υπεραξία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τη ε, υπηρεσία εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ήδη έχουν πετύχει την ισορροπία σε όλη την υπηρεσία μα, αλλά υπάρχουν ακόμα ανισορροπίε σε διάφορε υποκατηγορίε προσωπικού και τώρα αυτό εξετάζουμε. Εξετάζουμε τι ανισορροπίε, προσπαθούμε να τι ε, καλύψουμε. Ένα αυτό αφορά τη, από αυτά αφορά τη, τη διοίκηση. 46% των επικεφαλής αντιπροσωπείων ήταν διπλωμάτε των κρατών μελών το 2014 όταν έλαβα τα καθήκοντά μου. Τώρα είναι 43% μειώνεται αλλά ακόμα πιστεύω ότι ε, υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Ε, μπορούμε να πετύχουμε ε, καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη διοίκηση Πρέπει να πω ότι η ανισορροπία εντός της διοίκησης είναι αντίστροφη Λοιπόν, εντό του συστήματο γενικά έχουμε ισορροπία, αλλά υπάρχει ανισορροπία μεταξύ αντιπροσωπιών και κεντρική διοίκηση. και θα πρέπει να καλύψουμε τι ανισορροπίες, όποια κατεύθυνση και να έχουν αυτέ. Και εδώ κλείνω, λοιπόν, που μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να είμαι όσο δυνατόν πληρέστερη στην παρουσίασή μου. Γι' αυτό ζήτησα από τον Γενικό Γραμματέα να δημιουργήσει δύο task force, δύο ομάδε κρούση. Η μία θα εξετάζει το θέμα αυτό, ίσε ευκαιρίε και και ίσες ευκαιρίες για τα δύο φύλλα. Πέρσι τον Ιούλιο μας έδωσαν εκθέσεις οι δύο task forces και οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούν να εφαρμόσουν τις συστάσεις και τις βελτιώσεις που έχουν προταθεί. Από την task force πάνω από 100 μέλη του προσωπικού συμμετείχαν, άρα συμμετείχαν πάρα πολύ, ήταν ανοιχτή όλη η προσπάθεια και προφανώς είμαστε στη διάθεσή σας και ο Γενικός Γραμματέας μας σας δώσει λεπτομέρειες περί των διαφόρων μέτρων και των διαφόρων εφαρμοστικών μέτρων να κλείσω λέγοντα ότι η σημερινή μα ε, συζήτηση δεν αφορά μόνο θέματα προπολογισμού, αφορά την ενίσχυση του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωσης στον κόσμο και νομίζω γι' αυτό χρειάστηκα κάποιο χρόνο να το αναφέρω αυτό. Δεν έχουμε πολύ συχνά όμω τη δυνατότητα να ανταλλάσσουμε απόψει σε αυτή την επιτροπή. Ε, θεώρησα λοιπόν ότι είχα καθήκον πλευρά μου, ήταν ευθύνη δική μου να μοιραστώ μαζί σα τη γενική εικόνα δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Αν θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες μας και στους εταίρους μας ε, αυτά που περιμένουν από εμά, σε αυτή τη δεδομένη ιστορική στιγμή, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να είναι αποτελεσματικότερη δυνατή, θα πρέπει να έχει τους κατάλληλους πόρους να εργαστεί και το έργο σας πάντα μας βοηθούσε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και βασίζουμε στην υποστήριξή σας σε εποχές αυξανόμενων παγκοσμίων εντάσεων και αυξανόμενων προσδοκιών για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορείς να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Υπέχουμε ευθύνη ε, πρέπει να είμαστε αξιόπιστος, προβλέψιμος, συνεργάσιμος εταίρος ε, σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει και γι' αυτό θα πρέπει ο θεσμικό όργανο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να συνεργαστούν ο, κάθε φορέα με στα αυτονομία του ρόλου που έχει σαν ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και ξέρω ότι το Κοινοβούλιο πάντα συγχρονίζεται με αυτή την προ, ε, προσέγγιση. Σα ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Λοιπόν, είχαμε κάποιο χρόνο και γι' αυτό είχα την πολυτέλεια να μακρηγορήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ όπως γνωρίζετε. Εμείς δεν είμαστε μανιακοί <clears throat> σε εισαγωγικά τσιγκούνιδες, αλλά θέλουμε ακριβώς να μπορέσουμε μέσω των λαπανών μας να γίνουμε πιο γνωστοί και πιο ωφέλιμοι. <coughs> Θα ακούσουμε τον εισηγητή τώρα, ο οποίος έχει προετοιμάσει τις γραπτές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις σας ήταν πλήρης βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Χβάλη. <coughs> Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Αντιπρόεδρο για την παρουσίασή της και για τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο όπου δόθηκαν απαντήσεις σε συγκεκριμένα και ενδιαφέροντα θέματα τα οποία προκαλούν πάρα πολλές συζητήσεις. Ευχαριστώ και τον Πιέτρο Ρούσο για την παρουσίασή του και για τις πληροφορίες που έχει ήδη στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτήν την περίοδο διεθνούς αστάθειας έχουμε ανάγκη από μια υπηρεσία εξωτερικής δράσης ισχυρή και που προασπίζεται τις αξίες της Ένωσης και τις δημοκρατικές αξίες. Η απαλλαγή δεν περιορίζεται λοιπόν στην εξέταση μόνο διοικητικών λειτουργιών, αλλά και την προστιθέμενη αξία την οποία προσφέρει μέσω των ενεργειών που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια η υπηρεσία αυτή, και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη μετανάστευση και για την εμπορία ανθρωπίνων όντων και για θέματα λαθρεμπορίου, ναρκωτικών κτλ. Είναι θετικός ο ρόλος της υπηρεσίας λοιπόν εξωτερικής δράσης. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες βέβαια σε σχέση με τη διαχείριση του προϋπολογισμού. Καταρχάς οι διαδικασίες προμηθειών. Όπως είπε το ελεγκτικό συνεδρίο, οι αντιπροσωπείες έχουν κάποιες δυσκολίες στη διαχείριση των συστημάτων προηθειών. Ε, προβλέπονται από ό,τι διάβασα ε, διαδικασίες κατάρτισης και παρακολούθηση των ενεργειών τους. Κατανοώ ότι είναι δύσκολο για τις αντιπροσωπείες να διαχειριστούν τις διαδικασίες, αλλά απαιτείται να υπάρξει μεγαλύτερη και καλύτερη γνώση. Occorrono pratiche sane per evitare e Πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον λάθη και μη κανονικές εκτελέσεις του προϋπολογισμού, γιατί αυτό δημιουργεί κινδύνους απατών. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από την πλέον διαφανή τεκμηρίωση έτσι ώστε τα προγράμματα της ε, Επιτροπής να μην χαρακτηρίζονται, της υπηρεσίας μάλλον και των αντιπροσωπιών της να μην χαρακτηρίζονται μη κανονικά. Ιδιαίτερα στις αντιπροσωπίες όπου στο παρελθόν έχουν σημειωθεί κάποιες ε, μη κανονικές διαδικασίες. Ε, τώρα, έχουμε κάποιες ειδικέ ανησυχίες σε σχέση με το ότι 40% των δαπανών των αντιπροσωπιών είναι τα κτίρια. Το κόστος είναι υψηλό, είναι αναμενόμενο αυτό. Στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο λέγεται ότι θα χρησιμοποιήσετε εμπειρογνώμονες, αρχιτέκτονες και μηχανικούς για να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Πώς μπορούμε να εξετάσουμε ότι τα συμβάλλα... οι συμβάσεις αγοράς ή ενοικίασης μέχρι τώρα είναι συμβατές σε επίπεδο τιμολόγησης με τις τιμές της αγοράς και σε ποιο βαθμό μπορεί να υπάρξει αναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά όργανα να ξοδεύουν περισσότερο από όσο πρέπει. Η συνεργασία σας με την ΕΚΟ ε, θα μπορούσε να μειώσει ακόμα περισσότερο το κόστος λειτουργίας σας. Τώρα για την απλοποίηση γενικά του προϋπολογισμού. Εσείς κάνετε κάποιες προσπάθειες, ε, το κόστος ε, των αντιπροσωπιών καλύπτεται πλήρως από τον προϋπολογισμό σας. Ε, τι πιστεύετε μπορείτε να κάνετε περαιτέρω στα θέματα απλοποίησης για να γίνει ο προϋπολογισμός πιο διαφανής. Τώρα για τους σταζιέρ και γενικά ε, αυτοί οι οποίοι δεν αμείβονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης τους και θα πρέπει φυσικά να στηριχθούν και να καλυφθούν οι μισθολογικές τους ανάγκες. Θα πρέπει να μας ε, δώσετε κάποιες εξηγήσεις ε, και να μας πείτε τι συστάσεις έχουν γίνει από την διαμεσολαβήτρια. Τώρα για το κόστος των αντιπροσωπιών, αυτό είναι το πιο ακαθόδες θέμα. Στις εφημερίδες δημοσιεύθηκαν πολεμικά άρθρα για τις αντιπροσωπίες. Πέρα από το απλό θέμα του κόστους, το οποίο είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα είναι το πώς ζητείτε να καλυφθούν τα κόστη αυτά και πώς τελικά καλύπτονται. Μέχρι τώρα έχουν δημοσιοποιηθεί ε, τα στοιχεία του κόστους λειτουργίας των αντιπροσωπιών για τους δύο πρώτους μήνες του 2016. Θα πρέπει να συνεχίσετε να δημοσιεύετε τα στοιχεία αυτά για να έχουμε ακριβώς τεκμηριωμένα στοιχεία και εξοδακάλυψης ταξιδιών που καταλαβαίνω ότι είναι πολλές φορές απαραίτητα. Λοιπόν, θα αφήσω πάλι το λόγο ε, στο ελεγκτικό συνέδριο και στην ε, Αντιπρόεδρο έτσι ώστε να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, 40-45 λεπτά μόνο, οπότε θα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Αντιπρόεδρε, σας δίνω αμέσως το λόγο για κάποια από τα σημεία στα οποία αναφερθήκατε θα ζητήσω από το Γενικό Γραμματέα να συμπληρώσει. Είμαστε όλοι Ιταλοί και θα συνεχίσω στα αγγλικά για να μην νομίζουμε ότι είμαστε στην Ιταλική Βουλή εδώ μέσα. Υπάρχουν διοικητικά θέματα τα οποία τίθενται και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είμαι εδώ. Νομίζω όμως το ότι ε, προσπαθούμε να μην ξεχνάμε το γιατί είμαστε εδώ και πώς είμαστε εδώ, νομίζω είναι σημαντικό. Ε, είναι σημαντική η δουλειά την οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να ε, δώσουμε μάχη θα στραφώ στον Γενικό Γραμματέα και τους συνεργάτες τους για θέματα προϋπολογισμού να μας δώσουν έτσι μεγαλύτερες, περισσότερες μάλλον λεπτομέρειες για τις διαδικασίες προμηθειών, για την τεκμηρίωση και για τα κτίρια. Αν και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω κάτι γύρω από αυτά. Καταρχάς, τα γραφεία και οι κατοικίες. Είναι ένα δύσκολο θέμα, όχι μόνο για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά και για όλα τα υπουργεία, όλες τις διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Από τη μία έχουμε το καθήκον πρέπει να είμαστε λιτοί θα έλεγα. Από την άλλη είμαστε εκεί για να αντιπροσωπεύουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσημα. Ως εκ τούτου λοιπόν απαιτείται να έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο απαιτεί κάποιο κόστος ε, έτσι ώστε να είμαστε πραγματικά αντιπροσωπευτικοί της Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν πολυτέλεια γιατί δεν είναι χαρακτηριστικό της δικής μας πολιτικής ταυτότητας. Η φήμη μας ε, σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με υπέρογα επίπεδα πολυτέλειας. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, λυτοί, αλλά έχουμε ανάγκη από αίθουσε συναντήσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε μία κάποια τάση, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, άλλων υπηρεσιών που θέλουν να μοιράζονται τα γραφεία με την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Δράσης. Αυτό το ενθαρρύνω και εγώ γιατί βελτιώνει και την προστιθέμενη αξία και το κόστος, μειώνει το κόστος και όταν συγκατοικούμε με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες μερικές φορές δίνουμε μια ενιαία εικόνα και πιο ισχυρή συνεπώς της Ένωσης. Βλέπουμε ε, τον οίκο της Ευρώπης ουσιαστικά. Το κάνουμε πολλές φορές και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι θετικό. Αλλά αυτό μερικές φορές επηρεάζει βέβαια ε, τα πράγματα γιατί απαιτεί ε, μερικές φορές αναδιαρθρώσεις του τρόπου λειτουργίας κτλ. Για τα υπόλοιπα θέματα έχουμε υψηλό κόστος για διάφορες προσαρμογές ε, των συστάσεων, σαν παράδειγμα η πρόσβαση, η ορατότητα των γραφείων. Αυτό απαιτεί ε, δουλειά πολύ, έργα για να γίνουν ε, τα γραφεία, ε, τα, γραφεία μας συγγνώμη, προσβάσιμα εύκολα επίσης και για την εξοικονόμηση ενέργειας απαιτείται μία επένδυση για να βάλουμε σαν παράδειγμα ηλιακούς ηλιακούς πίνακες, αλλά παρόλα αυτά αυτό είναι κάτι που θα εξοικονομήσει χρήματα ε, στο μέλλον, ενώ θα επιβαρύνει μία πρώτη ε, χρονική περίοδο. Ένα άλλο θέμα που αφορά πάντα τα κτίρια και το νομίζω ότι καλό είναι να το εξαρτήσετε. Είπατε για την ΕΚΟ και τη συνεργασία μαζί της. Όπως είπα εμείς ενθαρρύνουμε τις υπηρεσίες αυτές να ενταχθούν στους χώρους μας και στα συστήματά μας και να δουλέψουμε μαζί. Υπάρχουν άλλα δύο επιπλέον στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι τώρα έχουμε πίνακες οι οποίοι συγκρίνουν όλες τις πιθανές επιλογές στο επίπεδο ε, ε, πινάκων, το οποίο δεν ήταν ε, διαθέσιμο στο παρελθόν. κάποιες από τις συνέπειες τις οικονομικές τις οποίες είμαι θα υποχρεωμένοι να καλύψουμε τώρα προέρχονται από ανηλυμένες υποχρεώσεις ε, από το παρελθόν πριν καν έρθω εγώ τουλάχιστον ε, στην υπηρεσία. Διαχειριζόμαστε 180 γραφεία και 140 κατοικίες όπως είπα, τα θέματα ασφαλείας επηρεάζουν ιδιαίτερα οικονομικά το κόστος διαχείρισης, αλλά και την ίδια την επιλογή των κτηρίων. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε να είμαστε σε περιοχές όπου είναι και άλλα κτίρια διπλωματικών αντιπροσωπιών, κυρίως των κρατών μελών. Και είναι σε περιοχές οι οποίες δεν είναι οι ευθυνότερες αλλά είναι και περιοχές οι οποίες καλύπτονται καλύτερα σε επίπεδο προστασίας και ασφαλείας. Το τελευταίο σημείο για τα κτίρια είναι ότι γενικά είμαι υπέρ του να αγοράζουμε κτίρια και όχι να ενοικιάζουμε. Αυτό σημαίνει ένα υψηλό κόστος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή αλλά είναι κάτι το οποίο μας εκθέτει πολύ λιγότερο στις διακυμάνσεις της αγοράς στο μέλλον. Είναι μια καλή επένδυση για τη διαχείριση των πόρων που έχουμε στην διάθεσή μας και μας διευκολύνει επίσης και στην συγκατοίκηση σε εισαγωγικά με άλλες υπηρεσίες. Φυσικά κάθε φορά πρέπει να είμαστε σε θέση να ελέγχουμε το ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές. Δεν είμαι εγώ που το κάνω αυτό, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με αυτά. Και αυτή είναι μια πολιτική η οποία στο παρελθόν δεν ήταν πάντα αυτή που ακολουθεί το. Όπως είπαμε, εμείς είμαστε σε επαφή με εμπειρογνώμονες, το είπατε κι εσείς, έτσι ώστε να διαχειριστούμε σε επίπεδο δημοσιονομικό με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα επίσημα κτίρια και κατοικίες. Δεν έχουμε πάντα βέβαια τους ανθρώπινους πόρους οι οποίοι θα μας συνοδεύσουν για να κάνουμε τις απαιτούμενες επιλογές. Αλλά εδώ ίσως στα διάφορα να μπορούμε να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία, ιδιαίτερα για τα θέματα των προμήθειών. Το κόστος των αντιπροσωπιών είπατε ότι είναι το πιο δύσκολο θέμα. Κοιτάξτε, διαφάνεια, ακόμα και αν μας εκθέτει εν πολλής, ε, ε, η πλήρης διαφάνεια είναι ο βασικός στόχος. Εγώ είχα ζητήσει από τις υπηρεσίες μου, προετοιμάζοντας τη συνάντηση αυτή, να δουν το κόστος και τις επενδύσεις που χρειάστηκαν ε, των δαπανών για τα ταξίδια των Υπουργών. Και δεν υπάρχει τίποτα το διαθέσιμο δημόσια σε σχέση με το κόστος ε, της υποδοχής των διεθνών αποστολών. Ε, Υπάρχουν προϋποθέσεις και απαιτήσει για θέματα διαφάνειας, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο υπουργού, αλλά και ε, άλλους επίσημους εκπροσώπους μιας χώρας, όπως πρόεδρο, πρωθυπουργό κτλ. Ε, θέλουμε λοιπόν να υπάρχει διαφάνεια, ακόμα και αν αυτό πολλές φορές οδηγεί σε παρερμηνίες. Καταρχάς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα χρήματα με σωστό τρόπο και παραγωγικό. Για να το κάνουμε αυτό, για μένα, όπως επίσης και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά, ο βασικός κανόνας είναι η ευθυνότερη δυνατή επιλογή, η οποία όμως να καλύπτει τις ανάγκες τις οποίες έχουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. σε λίγες εβδομάδες θα πρέπει θα πρέπει να είμαι το πρωί στο Κουβέιτ, ε, το απόγευμα στις Βρυξέλλες και την επομένη το πρωί στη Σόφια. Λοιπόν, εν πολλής προσπαθούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες να μην κοστίζουν και εν μέρη το πετυχαίνουμε. Αλλά για υπηρεσιακούς λόγους και λόγω της παρουσίας μου εδώ μερικές φορές απαιτεί να κάνουμε ταξιδιωτικές ρυθμίσεις οι οποίες σε επίπεδο ε, δρομολογίων αεροσκαφών δεν είναι διαθέσιμες και απαιτείται να ενοικιάζουμε πτυτικά μέσα και ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και οι περισσότερες διπλωματικές υπηρεσίες δεν έχουν δικό τους αεροπορικό στόλο. Υπάρχει λοιπόν σαφής ανάγκη ενοικίασης πτυτικών μέσων και εκεί προσπαθώ να ταξιδέψω με άλλους συναδέλφους, υπουργούς μερικές φορές, άλλες αντιπροσωπείες, υπουργούς, επιτρόπους και μοιράζουμε το κόστος. Για μία συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού ενός επιτρόπου μπορεί να είναι φθηνότερο το να χρησιμοποιήσει κανείς ένα δρομολόγιο αερογραμμών, αλλά από την άλλη μακροπρόθεσμα ο υπολογισμός και το τελικό κόστος ε, μπορεί να είναι υψηλότερο. Πάντως ε, ε, η ουσία είναι ότι εμείς επιδιώκουμε πάντα την ευθυνότερη λύση η οποία να μην επηρεάζει αρνητικά τη δουλειά την οποία πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα. Νομίζω ότι θα ήταν σωστό και οι εθνικές αρχές να ακολουθούν την ίδια αντίληψη για θέματα διαφάνειας, αλλά πάντως πρέπει να εξηγήσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να είναι ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά μέρη. Προσπαθώ να το πετύχω, σχεδόν το καταφέρνω, αλλά όχι απόλυτα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς ε, ε, είστε υπόλογοι γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις αποστολές τις οποίες είστε υποχρεωμένοι να αναλαμβάνετε. Για να μεταβαίνετε σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν ισχύει για όλους, για κάθε επίπεδο της διοίκησης θεσμό ή και πρόσωπο που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Υπάρχει καθήκον διαφάνειας και αναζήτησης ε, της καλύτερης δυνατής σχέσης τιμήματος και ωφελία. Είναι αναγκαίο αυτό, δηλαδή όπως λέγεται του αγαθού οικογένειά Η ίδια ε, σόφρον στάση. Η δαπάνη των χρημάτων πρέπει να γίνεται με διαφανή τρόπο και είναι απολύτως αιτιολογήσιμη. Γιατί, γιατί τότε και γιατί το συγκεκριμένο μέσον μεταφοράς. Αυτό όμω είναι πολύ σημαντικό γιατί μας επιτρέπει έτσι να εξηγήσουμε και το έργο μας. Θυμούμε την περίπτωση που αναφέρατε πριν, ήταν η πρώτη φορά δημοσίευση κόστου αποστολή όλων των επιτρόπων. Θέμα αυτό καθ' αυτό. Υπήρχε ένα θέμα σε μια αποστολή δική μου Αζερβαϊτζάν και Αρμενία. Υπήρχε πολιτικός λόγος που επέβαλε την επίσκεψη των δύο, των δύο αυτών χωρών, γιατί παίζουμε συγκεκριμένο ρόλο και είναι δύο σημαντικοί ανατολικοί εταίροι που έχουν θέματα μεταξύ τους και ήταν σημαντικό να μην επισκεφτούμε μονάχα τη μία πλευρά και την άλλη ταυτόχρονα και να αφιερώσουμε το ίδιο ποσόν χρόνου και στους δύο αυτούς εταίρους, το οποίο δεν είναι πάντοτε δυνατόν βέβαια ε, στη βάση των ε, δρομολογίων των εμπορικών ε, πτήσεων. Και ήταν και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο όμως, και διμερών σχέσεων, αλλά όχι μόνο, και τρόποι για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές. Αυτά συζητούνται δηλαδή. Έχει λοιπόν μια προστιθέμενη αξία να μπορώ να εξηγήσω τι είναι η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και σε τέτοιες χώρες που ηχούν κάπως εξωτικά τα ονόματά τους, ωστόσο είναι χώρες που έχουν και εντάσεις μεταξύ τους και χρειάζονται την ε, σύνδρομή μας αμφωτέρωθεν. Λυπούμε λοιπόν, μακρηγόρησα κάπως, αλλά ε, δεν είναι αμυντική η στάση μου. Αλλά γνωρίζω ότι και εσείς όλοι οι συναδελφοί μου έχετε καμιά φορά την ανάγκη, μάλλον υποχρώνεστε ορισμένε φορές να εξηγήσετε τα πράγματα αυτά. Νομίζω ότι ίσως ο Τζαν Μάρκο, ο συνεργάτης μου, θέλει να προσθέσει κάτι για τις προμήθειες και για... Και για τις απαντήσεις στις 53 ερωτήσεις σε αυτό το εξαντλητικό ερωτηματολόγιο. Ο εκπρόσωπος του... Ε, Έχω την εντύπωση ότι οι διάφορες αντιπροσωπείες έχουν τη διακριτική ευχέρεια να επιλέγουν κτίρια καθώς και διπλωματικές ε, ε, αξιοσημείωτες εξοικονομήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Για κτίρια. Κατοικίες και ε, αντιπροσωπείες σε άλλες χώρες. Ράστης. Παρακαλώ, εάν λόγω διαφανίας μας δώσετε λεπτομέρειες, πόσο περισσότερο χώρο χρειαζόταν διακομματική ομάδα, από την εμπειρία μου είδα ότι στα ανθρώπινα δικαιώματα και την εξηθρησκεία είναι τεράστια με αυτούς που συνομιλώ και αυτοί δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Και δεν έχουν κίνητρο. Έχετε κάποιον που έχει γνώσεις, κυρία το μεταξύ. Ο κ. Γιάφορο. Ο σκιώδης ηγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Μογκερίνη που ήρθε εδώ. Πες ήμουν εισηγητής για την απαλλαγή και θα θυμόσαστε ότι έπρεπε να συζητήσουμε πολλά σημαντικά θέματα. Είχαμε κάποιες αλλαγές και εξελίξεις, υπάρχουν και ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν φέτος. Πρώτον, δύσκολο θέμα, πολύ δύσκολο. Καμιά φορά υπάρχει λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ οικονομικής διπλωματίας, σημαντικός στόχος της διπλωματίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, και των ομάδων και των πιέσεων του lobbying η υπηρεσία εξωτερική δράση. τι μπορεί να κάνει για να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ οικονομική διπλωματίας και των λόμπι και τι εγγύησει υπάρχουν για το σαφή διαχωρισμό. Πρώτη ερώτηση αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Τα κονδύλια που στηρίζουν την υπηρεσία εξωτερική δράση. Είναι περιπλοκότατο το σύστημα, το ξέρουμε. Πολλά κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πέρα από τον προπολογισμό τη υπηρεσία εξωτερική δράση. Μπορεί να πλουστευτεί το σύστημα για τα κονδύλια που διατίθενται για την υπηρεσία εξωτερική δράσης. Οι λογαριασμοί να είναι πιο ξεκάθαροι. Να διατίθενται οι παρέτητοι πόροι με μία γραμμή του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί είναι δύσκολο να δούμε ποια είναι η προέλευση των χρημάτων, από ποιο κονδύλιο προέρχονται και πώς δαπανώνται. Άλλη ερώτηση. οι αντιπροσωπείες πώς λειτουργούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπηρεσίες της εξωτερικής δράσης συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς στους διαγωνισμούς και στι στις προμήθειες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ταυτόχρονα συμμορφώνονται καμιά φορά και με την ε, τοπική νομοθεσία που εκεί οι κανόνες δεν είναι διαφανείς όσον αφορά τι προμήθειες. Μήπως πρέπει να συμμετέχουν στην τοπική πραγματικότητα για τις προμήθειες, που ίσως εκεί να επικρατεί διαφθορά, να υπάρχει πολιτική μεροληψία. Τι εγγυήσεις υπάρχουν, ούτω ώστε να υπάρχει η σωστή διήθηση και να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες μας από τη διαφθορά. Και να γίνονται διαγωνισμοί εκεί με τρόπο που συμμορφώνονται με την νομοθεσία την τοπική και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία ερώτηση την περίπτωση το, του ξεπλήματος χρήματος ε, στο Αζερβαϊτζάν. και με τις περίεργες οικονομικές ροές των χρημάτων και πώς επηρεάζουν οι, ε, επηρεάζει το Αζερβαϊτζάν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το διελευκάνει αυτό. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε παρόμοιες τέτοιες περιπτώσεις και παρόμοιες απειλές στο μέλλον. Ευχαριστώ σκιώδης των φιλελευθέρων. Κύριε Κλίνς, έχετε το λόγο. Φορέστε να θέλετε τα ακουστικά σας, σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε κυρία, είπατε εκπρόσωπε στην αρχική σας τοποθέτηση ότι θέλετε να υποστηρίξετε και να υπερασπιστείτε τον πολυμερή χαρακτήρα των σχέσεων που αυτή τη στιγμή όντως απειλείται από τον τρόπο διαχείριση των θεμάτων από τον πρόεδρο Τραμπ. Θα ανέμενε κανείς οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπαραταχθούν καλύτερα και να ασκήσουν μια πιο συντονισμένη εξωτερική πολιτική. Πώς είναι ωστόσο δυνατόν παρόλα αυτά στην Γενική Συνέλευση της, ε, των Ηνωμένων Εθνών ορισμένε χώρες μέλη να κινούνται κατά, αντίθετα δηλαδή με την ε, Ευρωπαϊκή Γραμμή. Ο δε πρόεδρος ε, Τραμπ στα θέματα Ισραήλ και Παλαιστίνης έλαβε πρόσφατα απολύτως μονομερή θέση, δήλωσε δηλαδή ότι η Ιερουσαλήμ θα είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ και απειλεί ταυτόχρονα τις χώρες εκείνες μέλη του ΟΗΕ που δεν θα ψηφίσουν υπέρ του με οικονομικές κυρώσεις. Έχετε κάποιο σχέδιο για να διασφαλίσετε ώστε οι ανθρωπιστικές οι υποχρεώσεις απέναντι στους Παλαιστινίους θα συνεχίσουν να εκπληρώνονται. Παρόμοια είναι τα πράγματα με την Κούβα, όπου ο Ντόναλτ Τραμπ προσπαθεί να ανατρέψει την ε, πολιτική του προκατόχου του Ομπάμα. Αυτές τις ημέρες μάλιστα βλέπουμε ότι η Τουρκία παράνομα κατά βάση εισβάλλει στην Βόρεια Συρία και μάλιστα χρησιμοποιώντας γερμανικά όπλα και επιτίθεται κατά ομάδων, μπορεί να πει κανείς, Κούρδων, ότι είναι δηλαδή αμυγό Κούρδη. Εγώ αναμένω από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων κάποια τοποθέτηση, ωστόσο δεν έχω ακούσει τίποτα. Θέλω να ερωτήσω λοιπόν, πρέπει να αναμένουμε κάποια τοποθέτηση από την πλευρά της Επιτροπής Εξωτερικής ε, Δράσης και τι γίνεται με την δημοσιονομική διευκόλυνση που, με την μέσω της οποίας υποστηρίζει η Ευρώπη την Τουρκία για την υποδοχή σύρων προσφύγων. Τέλος, σχετικά με διεθνώς χρηματοδοτούμενα έργα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι όλοι οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε τέτοια χρηματοδότηση πρέπει να τηρούν τους ίδιους δημοσιονομικούς κανόνες. Τι εννοείται ακριβώς εδώ, πώς διασφαλίζεται ότι τα έργα εκείνα τα οποία θεωρεί άξια χρηματοδότησης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κρίνονται ομοίως και από άλλες διεθνείς οργανώσεις. Για το προσωπικό σας τέθηκαν ήδη ερωτήσεις. Εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός συνεργατών σας που όχι μόνο κάνουν πολλές υπερορίες, αλλά δεν παίρνουν καν την αδειά τους και την πληρώνονται. Πρόκειται για σύμπτωση ή έχει αναπτυχθεί ένα είδος νοοτροπίας που λέει κατά κάποιο τρόπο καλύτερα να δουλεύω παρά να βρίσκομαι σε άδεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Είναι εξής. Βελτιώσουμε την κατάσταση και να έχουμε σύντομες παρεμβάσεις ενό ή δύο λεπτών. E, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε, δεν έχουμε αρκετό χρόνο για μια σωστή συζήτηση και λυπούμε. Ίσως θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε άλλη μια συνάντηση μεταξύ μας. Έχω κάποιες ερωτήσεις που προετοίμασα και δεν θα μπορούσα στις όλες. Να πω εν συντομία τι θα ήθελα να μου πείτε. Πρώτα απ' όλα, η πολιτική ισότητας. Δεν αντιμετωπίζεται αρκετά σοβαρά. Αντίθετα με αυτά που είπατε, το 2017 από 43 άτομα που μπήκανε σε ε, θέσεις πρέσβεων, μόνο 12 ήταν γυναίκες. Και φαίνεται ότι δημιουργήσετε μία ομάδα, μία task force για τις ίσες ευκαιρίες. Θα ήθελα να ξέρω πόσα μέλη έχει αυτή η Task Force. Από τα μέλη της Task Force, πόσα, πόσες είναι οι γυναίκες. Άλλη ερώτηση. Η παρενόχληση των γυναικών. Είχαμε 75 υποθέσεις το 2017. 23 από αυτές εκκρεμούν. Υπήρξε αλλαγή τάσεων εν συγκρίση με την προηγούμενη τριετία. Εάν ναι, γιατί. Άλλη ερώτηση. Τι βοήθεια δώσατε σε θύματα παρενόχλησης. Άλλη ερώτηση. Γεωγραφική ισορροπία. Όσον αφορά μέλη αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Μόνο 15% των θέσεων ε, δόθηκαν στις 13 ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. στις χώρες που ήταν όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 13 μέλη. Όσον αφορά τις, ε, τον εφοδιασμό, τις προμήθειες. Καθορίζονται ποσά κάτω των 60.000 ευρώ ούτω ώστε να, υπάρχει, ε, να μην υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημοσίων προμηθειών. Κόστος συνεδριάσεων γιατί είναι πολύ πιο ακριβές οι συναντήσεις στις Βρυξέλλες από ότι εκτός Βρυξελών. 303 ευρώ ανά άτομο στις Βρυξέλλες, εκτός Βρυξελών 191 ευρώ ανά άτομο. Κάτι άλλο. Η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ενδιαφέρεται στο, για το πρόβλημα που αναφέρεται στο New York Times για τις πωλήσει όπλων στη Σαουδική Αραβία. Τι είπατε? Κοιτάξτε, τελευταία ερώτηση, υπόσχομαι τελευταία ερώτηση. Θα αφήσω όλες τις άλλες ερωτήσεις εκτός. Επέστρεψα μόλις από τη Χιλή. Στη Χιλή λοιπόν Έχουμε τρεις διπλωμάτες και μόνο στην αντιπροσωπεία μας εκεί. Και τώρα διεξάγονται δυσχερέστατες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Χιλής για εμπορική συμφωνία. Δεν είναι πολύ λίγοι. Τρεις. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της εν λόγω χώρας, της Χιλής και είπα είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος της Χιλής και υπάρχουν ε, πάρα πολλοί αντιπροσωποί του στη Χιλή. Η άποψή σας για αυτό το πρόβλημα ποια είναι. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια και μου δόθηκε, δεν μου δόθηκε αρκετό χρονικό διάστημα. Ο χρόνος είναι πρόβλημα, είναι περιορισμένος πόρος, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Να σας καλωσορίσω και εγώ, κυρία Μοντερίνη. Προέδρων των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπείων. Εκτιμώ την προσπάθεια την οποία κάνετε και θα ήθελα όμως να μπορέσουμε να συναντηθούμε και να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, σχετικά με κάποιες ερωτήσεις, θα ήθελα δύο μικρές ερωτήσεις στο οποίο θα πρέπει να βρίσκεται το προσωπικό της υπηρεσίας εξωτερικών σχέσεων. Γενικά η πλειοψηφία τους είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και εμεί φροντίσαμε και σαν Κοινοβούλιο και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να συμπληρωθεί κοντά στο επίπεδο το οποίο απαιτείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιο τρόπο μπορείτε να βελτιώσετε την επαγγελματικότητα Ε, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα ειδικά χαρακτηριστικά κάποιων ε, να Υπάρχει μια φορά το χρόνο όταν συναντώμεθα στις Βρυξέλλες, όταν έρχονται εδώ. Αυτό είναι κάτι το αρκετά αποτελεσματικό. Μήπως όμως θα μπορούσαμε να βρούμε και διαφορετικούς τρόπους έτσι ώστε να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας. Και τώρα για τη συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις όπως τα Ηνωμένα Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρχαν και προβλήματα σε σχέση με την αυτονομία της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη χρηματοδότησή της. Το θέμα είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την έλλειψη συντονισμού την οποία έχουμε μερικές φορές, κάποια ειδικά συστήματα για χώρες τις οποίες θα χαρακτήρισα κατά προτεραιότητα. Ε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ζητήσω συγκεκριμένη απάντηση, αλλά παρόλα αυτά Έχουμε δηλαδή ένα σωστό τρόπο επικοινωνίας έτσι ώστε όλες οι υπηρεσίες και όλα τα όργανα να μπορούν να επιλέγουν εν πάση περιπτώσει κάποιες περιπτώσεις κατά προτεραιότητα και να μην δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριος Καλώς όσον αφορά τη θέση αυτή. Δεύτερο σημείο. Σαν εισηγητή για του δημοσιονομικού κανονισμού, το θέτω το ερώτημα. Πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα. Και σα εύχομαι κάθε επιτυχία με αυτό. Ποια είναι η ανησυχία μου, τώρα που συντάσσω το δημοσιονομικό κανονισμό. Τα αποτελέσματα δεν είναι πάντα άριστα, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομή. Το πρόβλημα με τα καταπιστεύματα ποιο είναι, ότι μπλέκονται πολλοί φορεί και η συμμόρφωση και ο έλεγχο χείριση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεχόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Vždycky to beru tak, že je to příležitost ukázat, že stihnu svůj projev do dvou minut. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Πρώτα, οι δημόσιες προμήθειες. Αυτή είναι, αυτός είναι ο προβληματισμός μου. Δεν είναι κριτική αυτό που ασκώ. Καμιά φορά όμως είναι υπερβολικά περίπλοκα τα πράγματα, διότι εγκύπτουν οι ελεγκτές και στην τελευταίο κόμμα και τελεία. Ή έρχονται και εισάγουν όλο τον εξοπλισμό από την Ευρώπη. Ενώ είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να συζητηθούν που δεν μπορεί να τα λύσει το ελεγκτικό συνέδριο. Εμείς όμως ως ευρωβουλευτές όταν είμαστε καθοδόν και βλέπουμε ότι κάποιο εξοπλισμό έχει εισαχθεί από την ίδια την Ευρώπη. Εμεί θεωρούμε ότι αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Τώρα, δεύτερον, η ποιότητα του προσωπικού. Συμμετέσχουν σε αποστολή παρατήρησης εκλογών. Οφείλω να ομολογήσω ότι πολλές πληροφορίες μας έλειπαν. Δεν τις είχαμε από τους εκπροσώπους από τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως. Λάβαμε τις προφορίες αυτές από τους Αμερικανούς. Σχετικά δηλαδή με ε, τρομοκρατικές απόπειρες, επιθέσεις και διάφορα τέτοια. Και μάλιστα μια επίθεση που έγινε αμέσως μετά την αποχώρησή μας από ένα σημείο που είχαμε πάει να ασκήσουμε έλεγχο. Και άλλη απόπειρα έγινε ακριβώς πριν να φτάσουμε εκεί. Όμως εδώ μιλούμε για προσωπικό το οποίο πληρώνουμε εμείς. Αυτοί θα πρέπει να φροντίζουν για την ασφαλειά μας. Και τέλος, θα πρέπει να είναι κανείς ρεαλιστής. Μετά από το 2004 προσθέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές νέες χώρες μέλη. Εγώ ρώτησα πόσοι Τσέχοι, Ρουμάνοι, Πολωνοί συμμετέχουν στην ε, υπηρεσία σας και σε ποιες θέσεις. Και όταν κάνετε, όταν κάνετε διαγωνισμούς, τις θέσεις καταλαμβάνουν Ισπανοί, Πορτογάλοι, Ιταλοί κλπ. Ούτε Τσέχοι, ούτε Ρουμάνοι, ούτε Πολωνοί. Πώς τα βάλετε μέσα τις χώρες αυτές, αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ο κ. είναι ο τελευταίος. είναι σαν το είπατε σαν τον αγώνα ποδοσφαίρου και τώρα μιλάω τώρα σε, στην παράταση. Ίσως πρέπει να πετύχω το χρυσό γκολ και να τελειώσει η συνεδρίαση, σύμφωνα με την παροιμία Είμαι από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, κυρία Μογκερίνη. Είμαστε ουδέτερη χώρα. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Σε τέτοιο βαθμό που στη, συνθήκη της Λισαβ... στη δημοσίευση μας στη συνθήκη της Λισαβόνας εμείς καταψηφίσαμε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Για οποιοδήποτε λόγο διεξήχθη κι άλλο δημοψήφισμα διότι η Ευρώπη δεν πήρε την απάντηση που επιθυμούσε από το πρώτο δημοψήφισμα και στο δεύτερο δημοψήφισμα μα δόθηκαν διαβεβαιώσει όσον αφορά την ουδετερότητά μα και ότι δεν υπήρχε κάτι για το οποίο να ανησυχούμε. Στην Ιρλανδία είναι σαφέστατο ότι ίσω να μην είμαστε τόσο υπέρμαχοι εκείνων που υποστηρίζετε εσεί και άκουσα αρκετέ φορέ να λέτε και άλλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατείνονται ότι η κοινή πολιτική ασφαλείας και αμήνης μεταξύ 100 μερών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, την χάνει τεράστιας υποστήριξεις. Εγώ προβληματίστηκα όταν το άκουσα αυτό και είδα στοιχεία ξεχωριστά για τη δημοκρατία της Ιρλανδίας. Ζήτησα να μου δώσουν απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάτε για ανοιχτή προσέγγιση διαφάνεια. Δεν είδα απαντήσει. Οι απαντήσει που πήρα είναι αόριστε, δεν μου δίνουν λεπτομέρειε όσον αφορά συγκεκριμένη υπηρεσία για την Ιρλανδία αν υπάρχει Α, δεν ξέρω αν έγινε με, σε με, τον ίδιο τρόπο ότι κάτι με τη Ευρωπαϊκή Ενώσεις. Υποτίθεται ότι 1.300 άτομα εξέφρασαν την άποψή του στην Ιρλανδία και πιθανότατα μόνο 0% υποστήριξαν. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει τεράστια υποστήριξη ενδεχομένω. Θέλετε να επικρατεί διαφάνεια. Να είσαστε ανοιχτοί. μας δίνετε τα στοιχεία. Δεν μου αρέσει να ακούω ότι οι Ιρλανδοί πολίτες στην τεράστια πλειοψηφία θέλουν περισσότερη άμυνα και περισσότερες δαπάνες για πράγματα που καταστρέφουν τις ζωές των ανθρώπων ουσιαστικά. Μπορείτε να μου δώσετε στοιχεία. Φαίνεται ότι γίνονται δημοσκοπή σε αυτή τη φάση ούτω ώστε να φαίνεται καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλη δημοσκόπηση έγινε. Και με ερώτηση, θεωρείτε ότι είναι κάτι θετικό η ασφάλεια. Πώς το καλό βγήκε 100%. Μόνο 78%. Και τώρα λέτε ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα. Πρέπει να ανακατευθεί η Ιρλανδία στην Πέσκο κλπ. Με ενδιαφέρει πολύ η δουλειά που κάνετε. Παρακολουθώ αυτά που κάνετε. Προσπάθησα να μπω και να στην ετήσια συνεδρίαση της ε, υπηρεσία ε, εξωτερικής δράσης προσπάθησα να μπω και με έδιωξε η αστυνομία και ζήτησα γιατί ένας αξιωματικός ασφαλείας χτύπησε την κυρία που ήταν δίπλα μου στην προσπάθεια που κάναμε να μπούμε στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Κυρία Αντιπρόεδρε, βλέπετε πόσο δύσκολη είναι η κάλυψη ενός θέματος από 360 μοίρες. Έχουμε διερμηνία μέχρι τις 11. Και μετά η συνέχεια, θα συνεχίσετε στα Ιταλικά, λέει στην κυρία Μογκερίνη ο πρόεδρος. Κανένα πρόβλημα για μένα. Μπορώ να καλύψω Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά και λίγα Ισπανικά. Αλλά πρέπει σε 11 να είμαι αλλού. Πρέπει να τελειώσουμε λοιπόν. Σε χρονισμό Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τα δεδομένα του Ευρωβαρομέτρου αναεθνικότητα δεν τα έχω αυτά. Δεν είναι δουλειά μου αυτή, αλλά μπορώ να τα συγκεντρώσω και να τα συζητήσω μαζί σας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να κάνω κάτι τέτοιο. Για τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη τοπικά. Δεν έχουμε καμία δυσκολία, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πρόσφατα έγινε μια προσπάθεια συνεργασίας με όλες τις χώρες μέλη, τα αποτελέσματα ήταν θετικά και το βλέπω και εγώ όπου πηγαίνω βλέπω ότι οι αντιπροσωπείες μας έχουν ανάγκη για μεγάλους χώρους γιατί η ουσία της δουλειάς που κάνουμε δεν είναι μόνο να συναντώμεθα με τους ομολόγους μας στη συγκεκριμένη χώρα αλλά και με τους ε, εκπροσώπους των κατών μελών οπότε πολλές συχνά ε, συναντώνται οι εκπρόσωποι οι διπλωματικοί των 28 χωρών, όχι μόνο σε επίπεδο ε, πρέσβεων, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών συμβούλων, κοινοβουλευτικών υποθέσεων κτλ. Έχουμε μια μόνιμη δηλαδή προσπάθεια συντονισμού με τα κράτη-μέλη τοπικά. Και μπορώ να σας πω σαν παράδειγμα ότι σε σχέση με τους στόχους της αηφορίας και τις κλιματολογικές αλλαγές όλοι οι διαπραγματευτές, μας, διαπραγματευτές ε, ε, στα Ηνωμένα Έθνη δεν θα προχωρούσαν αν δεν συντονίζαμε τις 28 χώρες και δεν θα πετυχαίναμε να πετύχουμε ε, την προσπάθεια και το τελικό αποτέλεσμα στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν έγινε η δουλειά μόνο στη Νέα Υόρκη και στη Βόσινγκτον αλλά ρωτήσατε γιατί έχουμε μεγάλα γραφεία στη Νέα Υόρκη και τη Γενέβη. Αυτό γίνεται γιατί ο συντονιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Υόρκη και τη Γενέβη, τις δύο έδρες των Ηνωμένων Εθνών, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι διαφορετικές συνεδριάσεις συντονιστικές ταυτόχρονα, μερικές φορές πέντε φορές την ημέρα, όχι μόνο μία φορά την εβδομάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί πραγματικά πάρα πολλές συναντήσεις και αίθουσες αντίστοιχα. Εφόσον πρέπει να